κύριο Κανιέτε. Σας εύχομαι καλή επιστροφή στα σπίτια σας ή στα ξενοδοχεία σας. Διακόπτεται η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.